Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στην ε, ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την έκθεση Knights Utenbrook. Ποιο είναι υπέρ, Διανατάσιο χειρό παρακαλώ. Κατά, αποχέ. δεκτή. Έκθεση μούλτερ. Ψηφίζεται μια τροπολογία σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο,